συγχαρούμε. Περνάμε λοιπόν τώρα στι ψηφοφορίε. Έκθεση Μορέιρα για το τροποποιημένο καταστατικό στροκανονισμού για το καουτσούκ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Τέιλορ για τη λειτουργία και εφαρμογή εκτιμών δικαιωμάτων των ταξιδεύων αεροπορικά. Ψηφίζουμε ονομαστικά εδώ. Παρακαλώ, τη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση ΡΑΠΚΑΙ. Έτσι, περάσπιση τη βουλευτική το ε, του κυρίου Ντεμαζίστρη. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ονομαστική. Όχι. Όχι. Δεν είναι ονομαστική ψηφοφορία. Είναι διανατάσσος της χειρός. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερη έκθεση Ράπκαϊ για το ίδιο θέμα έτσι, παράσπιση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Ντεματζίστρης. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θέλετε το λόγο. Εγκρίνετε, εγκρίνετε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριος Ντάβιντ. Σας παρακαλώ αν μπορεί να έρθει ένας τεχνικός ε, γιατί το μηχάνημά μου δεν λειτουργεί. Πρόεδρος, περνάμε στην τρίτη έκθεση Ραπκάη. Για το ίδιο θέμα ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση Ραπκάη. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Εντάξει. Επαληθεύουμε έναρξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την τέταρτη έκθεση ΡΑΠΚΑΙ. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ταβάρης. Να δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Ταβάρης. Δεν ξέρω που είναι στην αίθουσα, δεν τον βλέπω. Ε, ναι, παρακαλώ κύριε ταβάρης σύντομα. Merci, Madame la Présidente. Dear colleagues, the legal act that we are adopting today deals with questions... Η νομοθετική πράξη που θα εγκρίνουμε έχει να κάνει ε, με θέματα ζωή και θανάτου για πολύ ευάλωτου ε, ανθρώπου, του πρόσφυγε ουσιαστικά και θα μπορούσα να είμαι χαρούμενο, Αλλά χρειάστηκαν δύο χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό τον συμβιβασμό. Έχουμε τη δικασία συναπόφαση, αλλά περί καμία συναπόφαση ε, δεν πρόκειται. Δεν είχαμε προθεσμία στην πρώτη ανάγκη. Ουσιαστικά είναι διαδικασία συν μη απόφαση, μη συναπόφασης. Αγαπητοί συνάδελφοι και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Αρκεί μια απλή οργανική συμφωνία. Ας σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία μη συναπόφασης. Ας βρούμε έναν αποτελεσματικό δίκαιο τρόπο να νομοθετούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ταβάρες. Δεν υπάρχει πρόταση απόρριψης ή τροπολογία. Επομένως εγκρίνεται η θέση του Συμβουλίου. Δυνάμει του άρθρου 74 του κανονισμού μας ε, θα υπογράψει την απόφαση αυτή ο Πρόεδρος. Αποκινούμε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου μέσα στο μεσημέρι σήμερα. Περνάμε τώρα στην έκθεση Μορέιρα. Έλεγχο εξαγωγών μεταφοράς μεσητείας διαμετακόμιση ειδών διπλής χρήσης. Δεν υπάρχει πρόταση απόρριψη ούτε κάποια τροπολογία. Επομένως κηρύσω εγκριθήσα την θέση του Συμβουλίου και περνάμε